23.00 έχει δημοσιευθεί η ημερησία διάταξη και είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λίγη εδώ η συνεδρίασή μας για απόψε. Εύχομαι καλό βράδυ και καλή επιστροφή σε όλους σας. Ευχαριστώ.